στη συνεδρίαση της 16 Απριλίου ήλεγξε την εντολή της κυρίας Τόρες Μαρτίνες και του κυρίου Τουρκάνου και πρότεινε ομόφωνα από τις 25 Μαρτίου 2015 και αντίστοιχα 2 Μαρτίου 2015 να ε, θεωρηθεί ότι είναι έγκυρη η εντολή τους. Εφόσον δεν έχετε μας, δεν έχετε αντίρρηση